Ja, schönen guten Morgen. Wir setzen unsere Sitzung von gestern fort und kommen. Καλημέρα σας. Συνεχίζουμε τη χθεσινή συνεδρίαση. Έχουμε να ε, διεξαγάγουμε μια ψηφοφορία όσον αφορά τις ρηπογόνε ε, ρηπογόνες εκπομπές από τα οχήματα. Είναι όλοι εδώ. Να δούμε, ε, κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, να δούμε ότι δεν έχουμε υπεράριθμους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 Και έτσι ξεκινάμε. Πρώτη ψηφοφορία, τροπολογία 21-23 μαζί, δύο τροπολογίες υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 3 και 5 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύω. 3 και 5. Δύσκολα βλέπω τα χέρια σας σε αυτήν την αίθουσα. Πέραση ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 20, 20 κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 24 και πάμε στην 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική. Μαζί με την τροπολογία 29 υπάρχουν αντιρρήσεις για την ε, προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 29 με προφορική μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η παριθμόν 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 38 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 39 υπέρ κατά. Υπέρ συγγνώμη. Κατά. Επαληθεύω. Δεν έχω καλή ορατότητα στην αίθουσα, παρακαλώ. Την 39. Επαληθεύουμε την τροπολογία 39. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Απερίφθη. 15 υπέρ 28. Κατά. Απερίφθη. Η 40 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43-44 μαζί. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Πάμε στην 47 κατευθείαν. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48. κατά αποχές ε, απερίφθη. 49 με προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία. Όχι. Μαζί λοιπόν 49, 50, 52 και προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι λοιπέ καταπίπτουν. Πάμε στι αιτιολογικέ σκέψει Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 13. Προσθήκη στη 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 καταπίπτει έχει γίνει δεκτή λοιπόν όχι ψηφίζουμε 16 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Ένα λεπτό. Πάμε στην αντιλογική σκέψη 7, προφορική τροπολογία, μαζί με την τροπολογία 19. Έχει κανείς αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε. Κατά αποχές, κρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει και πάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρασε ψηφοφορίες. Τώρα <coughs> πέρα ψηφοφορίας. 35 πέρα. 8 κατά. Μία αποχή. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Κυρία Λουκασένσκα δεν είναι εδώ. Να τη διαβιβάσετε τι ευχαριστήσει και τα συγχαρητήρια, παρακαλώ. Korridor können Sie natürlich sagen. Ja, klar. Und dass die Dokumente auch alle auslagen, verteilt wurden. Please may I ask you... Παρακαλώ όποιος δεν ενδιαφέρεται να μείνει στην αίθουσα να αποχωρήσει, να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πίεση χρόνου σήμερα. ich komme meine Besuchergruppe rein. Ich hoffe, die So, bevor wir zum nächsten Tagesordnungs gehen. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέλω να καλωσορίσω μια ομάδα 30 επισκεπτών της Επιτροπής από τη Γερμανία, της κυρίας Μάισνερ προσκεκλημένη. Καλώς ήρθατε. Und kommen zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Da begrüße ich recht herzlich Katrin Trautmann. Καλωσορίζω εδώ την κυρία Κατρίν Τροτσμάν που είναι συντονίστρια για τον ε, διάδρομο της Ανατολικής Βαλτικής με μεγάλη χαρά, για της ε, Βαλτικής μεγάλη χαρά την υποδεχόμαστε εδώ λοιπόν. Έχουμε 35 περίπου λεπτά για την παρουσίαση, αλλά ξέρετε, ούκεν το πολλό το F. Κυρία Τροτσμάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Ξέρω πως σήμερα γιορτάζετε τα γενέθλιά σας και ξέρω και πόσο σας ενδιαφέρει το σχέδιο για το τρένο υψηλής ταχύτητας προς τη Βαλτική και ελπίζω τα επόμενα γενέθλια να τα γιορτάσουμε μαζί με τα εγγένεια αυτής της γραμμής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποδέχεστε στην Επιτροπή σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που κινητοποιηθήκατε για να στηρίξετε τις προσπάθειες των συντονιστών για να προκρίνουν την χρηματοδότηση για ένα σχέδιο το οποίο σας παρουσιάζουμε εδώ. Φοβηθήκαμε πως το σχέδιο Juncker θα απορροφήσει πολλά από τα κονδύλια τα οποία εμείς χρειαζόμαστε και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να κάνω μια σύντομη παρουσίαση για να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του διαδρόμου αυτού. 3.200 χιλιόμετρα. Στο βορρά της Ευρώπης αποκλειστικά. Δεν υπάρχει σύνδεση λοιπόν μεταξύ των ε, θαλασσών στο βορρά της Ευρώπης και των υπολείπων θαλασσών όπως η Μεσόγειος. Τέσσερις χώρες από την Ευρωπαϊκή Δύση, τέσσερις χώρες που έγιναν μέλη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, Πολωνία, χώρες της Βαλτικής και αυτό αποδεικνύει τι διακυβεύεται είναι η ίδια η ισορροπία μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης αυτού του διαδρόμου, κάτι πολύ σημαντικό. 17 αστική κόμβη. Ξέρετε πως αυτή η αστική κόμβη είναι πολύ σημαντική, γιατί έχουν ε, το ρόλο του κόμβου για τα πόλη μέσα, κάτι το οποίο θα πρέπει να επιτελέσουν αποτελεσματικά γιατί έχουμε οδική, σιδηροδρομική και πλωτή σύνδεση. 16 αεροδρόμια, 32 εσωτερικοί λιμάνες, λιμάνες δηλαδή σε ε, ποταμούς και 13 από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, δηλαδή πύλη εσωτερική αγοράς. 17 ε, μεγάλη σιδηροδρομική σταθμή τέρμιναλ και 8 συνοριακά περάσματα. Άρα λοιπόν ε, πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν για να λειτουργήσει ο διάδρομος. Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα. Καταρχήν η ίδια συνοριακή διάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η ε, γραμμή ε, με τις σωστές διαστάσεις, ε, μάλλον με τις ίδιες διαστάσεις που να ενώνει τις χώρες Βαλτικής και την Πολωνία. Είναι διαφορετικό το πλάτος των γραμμών εκεί. Ένα πρόβλημα. Επίσης, ε, φορτία, εμπορευματοκιβώτια, εμπορικές σιδηροδρομικές διαδρομές. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, Έχουμε το πρόβλημα με το λιμάνι της, ε, του Μπρέμεν, όπως επίσης και με το Βερολίνο, που θέλουμε εκεί να ενώσουμε και σε σύνδεση με τις φλωτές δυνατότητες που έχουμε. Τρίτον, διαλειτουργικότητα. Ξέρω πως η Επιτροπή σας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Ο κύριος Λέβιν θα πάρει το λόγο μετά από μένα. Σε στενή συνεργασία με τον κύριο Βίνκ αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της ε, διαλειτουργικότητας και των ε, τριών συνοριακών ε, διασυνοριακών τμήματων που διαθέτουν αυτό το μηχανισμό ε, και συζητάμε για το πώς θα επεκτείνουμε αυτή τη δυνατότητα ναι. και σε άλλους που χρειάζονται αυτό το τεχνικό, τεχνολογικό μηχανισμό. Επίσης, αναλύσαμε με όλα τα στοιχεία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προσφέρουν τα διάφορα λιμάνια. Ένα από τα σημεία κλειδί για να πετύχει ο διάδρομος είναι τα θαλάσσια λιμάνια που επιτρέπουν τις μεγάλες συνδέσεις. Όχι μόνο Άμστερνταμ, Ρότερνταμ και Αμβέρσα, αλλά Αμβούργο και το ελεύθερο λιμάνι της Ρήγας, του Τάλιν. Η συνεργασία μεταξύ Τάλιν και Ελσίνκη σε επίπεδο ε, λιμανιών που είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα που επιτρέπει μέσω της υδροδρομικής σύνδεσης οι επιβάτες και τα εμπορεύματα να ταξιδεύουν ελεύθερα. Αυτά θα πρέπει να τα συμπληρώσουμε. Για τις πλωτές οδούς διακυβεύονται σημαντικά θέματα υποδομών. Έχουμε και γέφυρες αλλά και διόργες οι οποίες θα πρέπει να χτιστούν. Έχουμε σημεία συμφόρησης κοντά στα αστικά κέντρα. Και βέβαια το θέμα της ασφάλειας για το δίκτυο της Βαλτικής. Ενδεχομένως αυτό μπορούμε να το λύσουμε χρησιμοποιώντας κάποιες εναλλακτικές λύσεις για τα καύσιμα έχουμε και τα αεροδρόμια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και εκεί σύνδεση με ε, τις οδικές και σιδεροδρομικές μεταφορές. Επενδύσεις. 291 σχέδια επενδυτικά έχουν εντοπιστεί και χρειάζονται να υλοποιηθούν για να έχουμε αυτά που επιθυμούμε μέχρι το 2030 που έχουμε πει πλήρης εφαρμογή και λειτουργία. 122 είναι σιδηροδρομικά, 67 σχέδια είναι οδικά, 82 είναι λιμενικά και αφορούν και τις εσωτερικές ε, πλωτές οδούς και οι 20 σχέδια έχουν να κάνουν με αεροδρόμια. Για τα 291 αυτά σχέδια έχουμε υπολογίσει ένα απολογισμό 133 δις ευρώ σε τιμές του 2014. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες. έτσι ώστε να ορίσουμε μια ε, κατανομή των κονδυλίων η οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος της αξιολόγησης των σχεδίων που έχουν κατατεθεί για τους διάφορους διαδρόμους και στις 29 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει ποια έχει επιλέξει στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη. Ως συντονίστρια πρέπει να σας πω τι έκανα όλο αυτό το διάστημα. Ήρθαμε σε επαφή με όλους τους υπουργού συγκοινωνιών στα διάφορα κράτη-μέλη. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μία προσέγγιση, η οποία θα είναι ανοιχτή σε όλους, που θα φέρει όλους τους εταίρους κοντά, τις διοικήσεις, τις εθνικές, αλλά και παράλληλα τις περιφέρειες, τα αστικά κέντρα της πόλης, γιατί θεωρούμε πως για να πετύχει το σχέδιο αυτό θα πρέπει να στηριχθεί από όλους τους πολίτες. Γιατί είναι ένα τεράστιο project υποδομών. Είχαμε και δημιουργείς επαφές, επαφές με το μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που συνεχίζονται ακόμα και συμμετείχα και εγώ σε αρκετές περιφερειακές πρωτοβουλίες Έχουμε δημιουργήσει ένα βήμα στο οποίο θα εκπροσωπούνται ε, οι περιφέρειες που, ε, από τις οποίες περνάει ο διάδρομος και που θα συνεδριάσει κατά τις τέντη ημερίδες στη Ρήγα. Οι Ολλανδοί είπαν στην δική τους Προεδρία πως θα προωθήσουν το θέμα αυτό. Να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε και με τη βοήθεια των Φιλανδών και να δώσουμε ε, πολύ σημασία στο λογισμικό, στις τεχνολογίες επικοινωνίας και το τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο ε, ε, τεχνολογικό γενικότερα. Αυτό περιγράφει το ρόλο μου το τελευταίο διάστημα. Για το σχέδιο αυτό που είναι και μάλλον το εμβληματικό σχέδιο, την αυαρχίδα ε, του project που είναι το κομμάτι που αφορά τη συμφόρηση στις τρεις χώρες της Βαλτικής είπαμε πως θα επιλέξουμε κάποια σχέδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία ε, θα ε, υλοποιηθούν μέσω ενός κοινού σχήματος, το οποίο δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2004 ε, και που θα εκινήσει σε πρακτικό επίπεδο αυτά τα σχέδια. Άρα λοιπόν αυτό θα ενώσει όχι μόνο όσους συμμετέχουν σε αυτό το ε, joint venture, αλλά θα φέρει πιο κοντά και τις πολωνικές και τις λιθωνικές αρχές, οι οποίες έχουν ανάγκη να μια μεγαλύτερης προσέγγισης στο θέμα αυτό. Εγώ θα είμαι εκεί ως παρατηρήτρια και χαίρομαι που οι χώρες της Βαλτικής είπαν πως μέχρι το 2025 θα έχει λήξει ε, το έργο αυτό. Η ανακοίνωση θα σας παρουσιαστεί κατά τις επόμενες ημερίδες TNT. Για τις προτεραιότητες να σας πω τι θα συμβεί. Καταρχήν, για τις σιδηροδρόμους στις χώρες της Βαλτικής θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το κομμάτι αυτό από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλα τα κράτη-μέλη πως είναι το μοναδικό, ως το μοναδικό σχέδιο το οποίο ενώνει την ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και γι' αυτό θεωρούμε πως είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι θα ήθελα και εσεί να το φροντίσετε ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε. Έχουμε επίσης τα φράγματα του Άμστερνταμ που αποτελούν μια προτεραιότητα ε, για εμάς είπαν οι κατοχώρε που θα προσπαθούσαν να, βρίσκουν και ιδιωτικ... να βρουν και ιδιωτικά κονδύλια έτσι ώστε να μειωθεί η ανάγκη ε, μέσω του δικού ε, μηχανισμού να ε, χρηματοδοτηθούν. Για τα εσωτερικά λιμάνια και για την ένωση μεταξύ ε, πλωτών και σιδηροδρομικών οδών να σα πω πω αυτό αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα. Αυτό είναι λοιπόν η σύνδεση με την ενδοχώρα. Μετά έχουμε την διαλειτουργικότητα και για τα υφιστάμενα κομμάτια του δικτύου αλλά και για τα νέα τμήματα των υποδομών έτσι ώστε να είμαστε πιο αποδοτικοί. Κυρίως εδώ έχουμε εδώ τους αστικούς κόμβους που θα μπορούσαν να συνδέσουν κάποιους από τους διαδρόμους μεταξύ τους. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Επαναλαμβάνω, θα σας τα παρουσιάσουμε στη Ρήγα στις ημερίδες 10T και σίγουρα η δική σας η Επιτροπή ε, θα ακουστεί από τα κράτη-μέλη ε, στις μελλοντικές συζητήσεις που θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ και εγώ για την πολύ καλή έκθεση. Έχουμε μερικού συναδέλφου, Τέλιτσκα, Μάισνερ, Τσίλσεν, Σλοτόφσκι, Πίπερ και υποφαινόμενο. Και εσεί. Και εσεί. Ναι, έλεγα κι εγώ. Ζήλε, ματελή, καρέ ματελή. Ναι, και έχουμε πίεση χρόνου. Παρακαλώ, μισή λεπτό έκαστος. Πάβελ Τελίτσκα. Καλημέρα. Πρώτα πρώτα, Πρόεδρε, να πω χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σας. Και βέβαια το πιο σωστό είναι, ως κάνουν gentlemen, να προσφέρετε μια σαμπάνια, αλλά αργότερα, το απόγευμα. Πολύ πλήρη ήταν αυτή η παρουσίαση. Πρόκειται για ένα έργο περίπλοκο. Έχει διαστάσεις που δεν τις έχουν τα παρόμοια έργα. Πάρα πολύ ξεκάθαρα μας τα είπατε και θα πάτε φαντάζομαι στο συμπόσιο αυτό της Ρήγας για τις ημερίδες των Ευρωπαϊκών Δικτύων και οι προσδοκίε είναι αυξημένε σε σχέση με τους στόχου που έχουμε. Εντάξει, και εσείς κατά τη θητεία σα. έξι μήνες, ένα χρόνο που ασχοληθήκατε πέστε μας κάποια πολιτική αξιολόγηση για πέστε μας για τις επιδόσεις του κάθε κράτους μέλους Ε, ό,τι και να κάνετε δεν μπορείτε να υποκαταστήσετε τα κράτη-μέλη για να κάνετε αυτό που θα πρέπει να κάνουν εκείνα. Κάποια κράτη-μέλη έχουν καθυστερήσει πολύ. Μιλάμε για 130 δις και πολλές φορές χάνονται τα κονδύλια του Connecting Europe. Άρα θα πρέπει κανείς να αποδώσει, θα πρέπει κανείς να κάνει το μερτικό του, ας πούμε, το ότι το αναλογεί ε, και αν δεν το κάνει, χάνει και τα χρήματα και τελείσει η ομοιρία και η όμορη χώρα, το, ο γείτονα το project. Άρα, τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη ε, ή τι δεν κάνουν, ούτως ώστε να κάνουν αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Κύριε Τχοτμάν, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τι είπατε για τη Γερμανία, τα γνωρίζω πολύ καλά. Είναι όλα από τη δική μου εκλογική περιφέρεια. Ε, το κομμάτι ύψιλον όμως του διαδρόμου ε, στη πλευρά της Βαλτικής δεν έχει περιληφθεί. Το, κανάλι της, ε, το παράκτιο κανάλι βλέπω με χαρά ότι παραμένει. Συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα. Σε ποιο βαθμό συμμετέχετε σε ε, συνεδριάσεις για τα Sea Basin Strategies για τη Βόρεια, για τη Βαλτική θάλασσα, γιατί πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι πάντα παρούσα η συντονίστρια ή ο συντονιστής θεωρώ. Αυτό θέλω να ρωτήσω, πόσο συχνά είστε παρούσα. Επίσης, ναι και αναφερθήκατε συγκεκριμένα έργα για το Αμβούργο. Έχουμε αρκετή ε, στενότητα χώρου εκεί. Είναι γνωστό, υπάρχει κάποια διάθεση ή σχέδιο για τη διεύρυνση του, ε, των δυνατοτήτων λιμενισμού από το σχέδιο The Juncker. Είπαμε, ακούσαμε αυτά που είπατε για τους ατοκφράχτες του Άμστερνταμ όπου θέλουν οι Ολλανδοί να προσελκύσουν ειδικούς, ε, ιδιώτες ε, επενδυτές. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να εγγραφεί στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker. Ευχαριστώ Νίλσον. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο ερωτήσει. Οι οποίε δεν έχουν τόσο πολύ να κάνουν με χρήμα, αλλά με διαδικασίε. Εσείς ως πρώην Δήμαρχο, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνομιλεί όχι μόνο με κυβερνήσει, αλλά και με τοπικές και περιφερειακές αρχές οι οποίες πρέπει να προσκαλεί σε συνεργασία το κράτος λοιπόν ή οι τοπικές αρχές βλέπετε να αναλαμβάνουν και να επιτελούν ο καθένας το μερίδιο του έργου που το αναλογεί. Επίσης, ε, σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη, τη Σουηδία, τη Φιλανδία, ε, σε τι θέση νομίζετε ότι βρίσκονται οι χώρες αυτές εάν αυτό το οποίο μας περιγράφεται τώρα ονομάζεται Βόρεια Ευρώπη ή Βόρειος Άξονας. Υπάρχουν πολλοί λιμένες ε, και στη Σουηδία που προσπαθούν να και διευκολύνουν πιστεύω την κίνηση μεταξύ Βορρά και Νότου. Ε, ποια είναι η θέση τους. Ευχαριστώ κύριε Σλοτόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, εύχομαι και εγώ χρόνια πολλά πρόεδρε επί τη ευκαιρία για την σας. Για την παρουσίαση. Έχω μια ερώτηση ε, έχω την ότι δεν άκουσα να λέτε τίποτα για τα πολωνικά σύνορα, Κτάνσβιν, Κουίσκα και άλλα. Τι θέση βλέπετε λοιπόν για τους ε, πολωνικούς λιμένες εκεί. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κύριος Πίπερ. Ε, ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Στατικών Επενδύσεων, το ΕΣΥ. Ακούσαμε πολλά έργα για υδατοφράχτες, ε, υδάτινες οδούς, σιδηροδρόμους. Κύριε Τροτμάν, πιστεύετε όντως ότι μπορείτε να, να βρείτε ιδιώτες επενδυτές για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Θεωρείτε πράγματι ότι το σχέδιο Juncker μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα για να προαχθούν αυτοί, οι άξονες των μεταφορών που εμείς με τόσο κόπο έχουμε συντηρήσει και προβάλλει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης η διασύνδεση μεταξύ κάτω χωρών και Ανατολικής Ευρώπης. Στις, ε, στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας κάτω χωρών μας λείπουν από τις ναι, πλωτές οδούς 20 μόλις χιλιόμετρα από τα κανάλια αυτό θα διευκόλυνε κατά τουλάχιστον μισή ώρα, μισή ημέρα ε, κέρδος χρόνου την μετάβαση από την περιοχή των κάτω χωρών προς την Ανατολική Ευρώπη. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν και γιατί να μην ε, φτιαχτεί αυτό το κομμάτι που λείπει ώστε να προσφέρουμε και για τις επόμενες γενναίες τη δυνατότητα για τις μεταφορές. Δεν μπορείτε να επηρεάσετε το σχεδιασμό των επιμέρους κρατών. Ευχαριστώ. Βίρκουνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε για την ε, εισηγήση, ευχαριστούμε για τις ε, προτάσεις. Ε, πολλές από τις προτάσεις με βρίσκουν σύμφωνος. Εγώ είμαι Φιλανδέζα, ε, άκουσα και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριο Νίλσεν, ο οποίο είναι Σουηδό, γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο διάδρομος ε, συνδέει την Ευρώπη με την ε, Βαλτική και θεωρώ ότι έτσι θα αναβαθμιστεί η περιοχή της Βαλτικής ακριβώς γιατί θα συνδεθεί με την Ευρώπη και από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι θα ωφεληθούν και τα αεροδρόμια στη Φιλανδία, μια που θα μπορούμε να έχουμε και πτήσεις τώρα από Ασία κλπ. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα ε, στην Βαλτική. Έχουμε πάρα πολύ αυστηρά όρια εκπομπής θείου και έχουμε και τους τερματικούς σταθμούς του φυσικού αερίου. Είναι σημαντικό το να υπάρχει ε, σύνδεση μεταξύ λιμένων και των αξώνων ε, οδικών μεταφορών. Νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσει το πράγμα ακόμα καλύτερα και θα πρέπει να βρεθούν κάποιες ε, λύσεις αλλά υπάρχει πρόβλημα τώρα ε, όσον αφορά τις συνδρομικέ μεταφορές στην περιοχή της ε, Βαλτικής. Είναι πάντως πολύ σημαντικό αυτό το έργο για την περιφέρεια εκείνη και θα ήθελα να μας πείτε αγαπητοί σε λεπτομέρειες την απόψη σας τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ Σίλε. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man arī priekšēt redzēt faktiski divus koordinātors. Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα. Βλέπω εδώ δύο συντονιστές. Τον κύριο Τέλτσκα. Και θα συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Τέλτσκα με πολύ οικοδομητικό τρόπο σε σχέση με την ε, Βαλτική. Όταν άρχισα εγώ τη δουλειά του συντοπιστή, ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι είδου εμπόδια βλέπετε να υπάρχουν ως προς την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου για το σιδηρόδρομο στη Βαλτική. Μιλήστε και με διπλωματικό τρόπο θέλετε, αλλά μιλήστε και περίφραστα καλύτερα. Και επίση θεωρώ ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα του χρόνου πρόκειται να διατεθεί σε κυκλοφορία ένα κομμάτι του σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Λετωνία και Πολωνίας από το Ταμείο Συνοχή, το οποίο όμω το κομμάτι αυτό δεν επιτρέπει τρένα υψηλής ταχύτητας. Εάν χρειαστεί λοιπόν να φτιάξουμε μια άλλη γραμμή δίπλα, τι έχουμε επιτύχει σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ευχαριστώ, Καραμαντελή. Ευχαριστώ πολύ, Κατρίνη Τροτμάνη, για την ε, παρουσίαση. Θα είμαι σύντομη και η πρώτη με ερώτηση είναι μήπως μπορείτε σήμερα να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για το πώς έχετε προσπαθήσει να εμπλέξετε τους ε, πολίτες ε, σε αυτό το έργο συνοσμού που έχετε αναλάβει. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Επίσης, είχατε συναντήσει κάποιες δυσκολίες και ποιες ήταν αυτές. Και η τελευταία ερώτηση. Πεςτε μας. Τι γίνεται με τον διάδρομο και το ΕΡΤΕΣ όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά τα υλικά. Υπάρχει ουσιαστική πρόοδος. Μήπως υπάρχει εμπλοκή και αν υπάρχει κάποιος εμπλοκή στην κατάσταση πώς προκαλείται. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ δύο λόγια. Έχουμε δύο στιγμές, λοιπόν και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυτή η γραμμή ευρωπαϊκή. Αλλά από το Λίστοκ ε, περνάει στο ΕΛΚ, στο Βάλκινα Κάουνας ή από την άλλη γραμμή την παραδοσιακή και έχουμε καταλήξει τελικά κάπου. Λέγεται ότι θα είναι σε δύο χρόνια έτοιμο το κομμάτι αυτό, μέσω του Ριστόκ προς τα σύνορα, πέραν των σύνορων. Και εδώ θα συμφωνήσω με τον Ρομπετσίλο ότι ουσιαστικά ε, σπαταλάμε χρήματα. Εάν φτιάχνουμε μία γραμμή η οποία δεν εξυπηρετεί την υψηλή ταχύτητα εμείς στη Γερμανία έχουμε ε, γραμμές υψηλής ταχύτητας που καλύπτουν και την τοπική και την περιφερειακή κίνηση, αλλά και την υψηλή ταχύτητα Φερρυπίν μεταξύ Βερολίνου και Αμβούργου. Υπάρχει, είναι δυνατόν και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια στοχευμένη προσπάθεια. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι σε αυτό. Ευχαριστώ κατά τα άλλα για την παρουσίασή σας. Έχετε το λόγο τώρα για να απαντήσετε. Τρότμαν, ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω όσο γίνεται σαφέστερα σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο. Ευχαριστώ τον Παύλ Τέρισκα γιατί είναι ο πρώτος βουλευτής ο οποίος ε, έθεσε ερώτηση και πρόκειται για κάποιον που έχει ε, γνώσεις ειδικέ στο τομέα. Έχει επιτελέσει σημαντικό έργο με τον ε, James που είναι εδώ πίσω και επίσης η Βέρα Κίσλερ παρακαθήμενη που είναι η σύμβουλός μου ε, στην Επιτροπή. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το, είμαστε αυτό το δίδυμα από γυναίκες και αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε σε σχέση με το διάδρομο. Τώρα, επίσης, ε, και για σας και πρόεδρε και για τον κύριο Ζήλ και για τους άλλους ε, βουλευτές θα πρέπει να σας, να σας πω για την ε, πολιτική αξιολόγηση μπορεί να γίνει, για το τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά τη στάση των κρατών μελών. Η πρώτη δυσκολία για όλου του διαδρόμου, αλλά και για τον συγκεκριμένο, είναι το ότι όλοι, όλοι ε, θέλουν ε, διάδρομο και θέλουν ε, να αντιπροσφέρουν ταυτόχρονα το, το, το αμοιβαίο και το συλλογικό συμφέρον. Επομένως, Πρόεδρε, το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο επίση επισημάνετε μεταξύ Κάνος και Μπιάλιστοκ. Μεταξύ δηλαδή Πολωνίας και Λιθουανίας. Και γι' αυτό το λόγο καθ' όλη αυτή την τελευταία περίοδο έχω πασχίσει πρώτα-πρώτα να φέρω μια προσέγγιση των απόψεων, να συμβαστεί η Πολωνία με την Λιθουανία, ούτως ώστε να απεμπλακεί όλο αυτό το, το, έργο που αφορά το σιδηρόδρομο εκεί, στη Βαλτική. Γιατί πρόκειται για μια συνολική γραμμή υψηλής ε, ταχύτητας Τρει βαλτικέ χώρε και συνδέεται με το υπόλοιπο δίκτυο μέσω τη Πολωνία. Χωρί αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για αποτελεσματικό δίκτυο. Είναι θέμα πολιτικό και γεωστρατηγικό και αφορά όχι μόνο τι τρει βαλτικέ χώρε και την Πολωνία, αφορά και την Φιλανδία που υποστηρίζει την πρόταση η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί στη Ρήγα. Οπότε Φιλανδία Πολωνία είναι παρατηρητέ σε αυτή την κοινοπραξία και ήδη είναι ε, παρατηρητές στην Task Force. Οπότε ελπίζουμε από εκεί και πέρα να υπάρξει μια κοινή διαχείριση. Και η DG Move επί τόπου πρόκειται να έχει επαφές με αυτούς τους δύο εταίρους μας για το σύνολο αυτής της γραμμής από Βαρσοβία μέχρι Κάουνας ούτως ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τις μελέτες των ε, Πολωνών που μας έχουν διαβαστεί για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα για το περιβάλλον, πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε, ε, πού μπορούμε να έχουμε καινούργιες γραμμές. Ε, έχουμε ταχύτητα ε, συνεχή 160 χιλιόμετρων την ώρα για να δούμε πώς θα γίνουν οι επενδύσεις στις χώρες της Βαλτικής. Στην περίπτωση τώρα της Λιθουανίας και εκεί θα πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά τις νέες γραμμές και ακριβώς με αυτή την κοινή προσπάθεια θα πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα γιατί για μένα ε, ο πρόκειται στρατηγικό, πολιτικό ε, όμως καταρχήν υπάρχει η καλή διάθεση, υπάρχουν και προβλήματα αλλά από πλευρά της πολωνικής κυβέρνησης υπάρχει αυτή η καλή θετική διάθεση και επίσης ε, από τη Λιθουανία υπάρχει δηλαδή ο έρωτας αλλά χρειάζεται η απόδειξη του ότι υπάρχει αυτή η θετική διάθεση. Υπάρχει διάθεση συμβασμού αλλά ο καθένας θέλει εγγυήσεις από τον άλλο. Άρα θα συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκομένους. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά την Βαλτική και το Σιδηρόδρομο που είναι η μας ε, τη σήμερα ημέρα. Διότι εκεί έχουμε τις πολιτικές δυσκολίες αλλά μας προστρίζει η κυβέρνηση της Γερμανίας, του Βελγίου, των κάτω χωρών και όλε όλες οι δυτικές χώρες έχουν καταλάβει τη σημασία του να ε, ολοκληρωθεί αυτό το έργο υποδομή Τώρα, όσον αφορά την κάτω Σαξονία, στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη προσπαθούμε να επιλύσουμε κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν τον ορισμό του διαδρόμου ας πούμε να ληφθεί υπόψη ο Έλβας και επίση τα προβλήματα του ποταμού Όντερ. Και γι' αυτό και τα λέμε όλοι οι εμπλεκόμενοι και τον Πατ Κόξ επίσης προσπαθούμε να συνδυαστούμε για τον διάδρομο της Σουηδίας γιατί δεν αρκεί μόνο το Ελσίνκι να εμπλακεί. Βέβαια, για τη Φιλανδία να δούμε αν θα καλύψουμε και τις φιλανδικές λίμνες που είναι ε, πλωτός ε, ε, διάδρομος και έχουμε επίσης και το κανάλι του Κιέλο ούτως ώστε να ενώσουμε τη Βόρειο Θάλασσα με τη Βαλτική τα λιμάνια από τη μία και από την άλλη γιατί πρόκειται για πριορισμούς, δηλαδή θέλουμε να, να, να, να κλείσει ας πούμε αυτό το κύκλωμα με αυτό το κανάλι. Améliorer euh, le, euh, euh le, la régulation, le règlement euh, lorsque il. Οπότε έτσι να γίνει κάποιο είδου ρύθμιση, να αναθεωρηθεί ο κανονισμό και επίση να δούμε τι θα γίνει με τα σημεία απόφραξη ε, και τι θα γίνει με του αστικού κόμβου. Έχουν εμπλακεί βεβαίως και οι τοπικές αρχές, συναντήσεις. Έχουμε το Ρέγγιο για Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία. Έχουμε το, την ε, Σάξ έχουμε το Βερολίνο κλπ. Οπότε έτσι έχουμε κινητοποίησει όλες τις επιμέρους περιφέρειες και είμαστε και σε επαφή με τις πολωνικές αρχές και υπάρχει μια ιδιαίτερη περιφερειακή διάσταση εκεί στην Πολωνία που θα επηρεάσει τη συνέχεια της πορείας μας. Υπάρχει το φόρουμ στην Ρήγα, φόρουμ των περιφερειών, θα γίνει άλλο φόρουμ περί το τέλη του έτους και για μένα είναι μια προτεραιότητα να συνεργαστώ εκεί και να έχουμε την τελευταία φάση αυτού του προγράμματος σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Τώρα όσον αφορά τον βορρά της Ευρώπης συμφωνώ 100% για το ότι δεν αρκούν αυτά όσον αφορά τις ε, πρώτες ε, ύλες και επίσης τις, ε, τα βασικά θέματα των μεταφόρων. Τα είπαμε τον Πατ Κόξ, τον διάδρομο Σκανδιναβία Μεσόγειος, οπότε να δούμε το πώς θα μπορούμε τελικά να έχουμε ένα τέτοιο όραμα, μια τέτοια οπτική για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα θα επισκεφθώ τον ε, οργανισμό ε, εποπτείας, ε, την κανονιστική αρχή Φιλανδίας και Βαλτικής. Να δούμε και τι μεταστάσεις υπάρχουν. Επίσης να δούμε τι γίνεται στους σιδηροδρόμους, τους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Φιλανδία, τα συστήματα μεταφοράς. Μια βελτίωση η οποία έχει ξεκινήσει Οπότε η συνεργασία εκεί είναι πάρα πολύ θετική και αυτό μου δίνει κουράγιο. Τώρα όσον αφορά τις στατικές επενδύσεις και το σχέδιο Juncker και εδώ εμπλέκεται η υπόθεση αυτή και δηλαδή και στο διάδρομο έχουμε το λιμάνι του Αμβούργου κάποιες διασυνδέσεις έχουμε τα, τους υδατοφράκτες στο κανάλι του Τβέντε και όλα αυτά θα τα προσέξουμε ξεχωριστά. Βλέπετε επομένω ότι υπάρχουν κάποια έργα τα οποία ξεχωρίζουν. Υπάρχει προσθέμενη αξία επομένω από οικονομική πλευρά. Αυτό και πρόκειται να αναδείξουμε. Τώρα κάποια άλλα ζητήματα για αεροδρόμια και για το κατά πόσον μπορούμε να έχουμε συνδρομικές συνδέσεις είτε για εμπορικά τρένα είτε για επιβατικά προς και από τα αεροδρόμια σε σχέση με το Ελσίνκι που είναι πολύ σημαντικό. Εκεί η συντονίστρια προσπαθεί να υποστηρίξει αλλά και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα κριτήρια που ισχύουν για τον διάδρομο. Και εδώ επομένως θα πρέπει πολλά να κάνουμε όσον αφορά τον αστικό κόμβο και τις βελτιώσεις. Ποια είναι σήμερα τα προβλήματα. Πολιτικά είναι και οικονομικά. Άρα θα πρέπει να γίνει προγραμματισμός που να επιτρέπει την υλοποίησή μας ε, στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών. Γιατί πολλοί λένε ναι, ναι, να γίνει η αρχή και βλέπουμε στη συνέχεια. Όχι, έτσι έγινε, έγινε αναμέτρηση δυνάμεων και παράθεση με αυτούς. Οπότε έτσι θα πρέπει να εμπλακεί και ο πολιτή, να υπάρχει επικοινωνία και αυτό θα βοηθήσει να αρθούν αυτοί οι φραγμοί. Και ο Παύλ Τέλιτσκα, πριν από μένα σαν συντονιστής, βοήθησε να υπάρχει επικοινωνία από πλευράς ε, κομισιών και από πλευράς κρατών μελών που θα διεξαγάγουν ε, τα έργα. Άρα να εμπλαγεί ο κόσμος. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση προς τα εθνικά κοινοβούλια, προς τον κόσμο. Κάποιες κυβερνήσεις ξεκάθαρα το είπαν. Θέλουμε τη βοήθειά σα. Και εγώ θα δώσω τη βοηθειά μου χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήμουν δήμαρχος και ξέρω τι γίνεται με αυτά τα μεγάλα έργα ε, αυτό, είχαμε αυτό το ΤΖΒ σε τρεις περιφέρειες της Γαλλίας ε, και είχε εμπλακεί τότε κάθε οικοδιαμέρισμα, κάθε πόλη κλπ. ούτως ώστε να αποδεχθεί ο κόσμος τη χρηματοδότηση αυτής της ε, υποδομής. Και να αποδεχθεί βέβαια φόρους, χαράτσια κλπ. <clears throat> Και όλα αυτά πήγαν πάρα πολύ καλά στη Γαλλία, επομένω μπορούν να γίνουν και σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα πρέπει πάντως να αποδείξουμε ότι χρησιμοποιούνται σωστά τα χρήματα και πάνε εκεί που πρέπει. Οπότε και έχουμε καλέσει όλους τους εταίρους, ε, λιμενικές αρχές, τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις, ούτω ώστε να υπάρξει μια επικοινωνία για το σχέδιο Γιούγκερ, για άλλα έργα, ας πούμε για το σιδηρόδρομο στις βαλτικές χώρες, αλλά ε, εκεί καλύπτει το σχέδιο Γιούγκερ, αλλού χρειάζεται συγκριματοδότηση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένα θεματολόγιο, ένα σχέδιο δράσης για να γίνουν όλα αυτά το 16. Πιστεύω πρώτα ότι θα, θα ξεπεράσουμε δυσκολίες. Ευχαριστούμε και σας για την υποστήριξή σας να το κάνετε αυτό στη χώρα σας. Αλλά σα διαβεβαιώ ότι αυτό ο διάδρομο και ο σιδηρόδρομος στη Βαλτική θα πρέπει για μα να είναι μέσα στι κορυφές έξι προτεραιότητε για αυτήν την ε, περίοδο όταν μιλούμε για, για το δίκτυο των ευρωπαϊκών διαδρόμων. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Κατρίν Τροκμάν. Και εμεί είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζω θα ήμασταν εδώ. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε στις προθεσμίες. Δύο σύντομες ερωτήσεις βλέπω, κυρία Μάισνερ. Πολύ γρήγορα, κυρία Τροτμάν. Δεν μου απαντήσατε. Θα συμμετάσχετε σε συζητήσεις για τη στρατηγική, για τη Βόρεια Θάλασσα ή για τη Βαλτική. Βλέπω ότι βαίνουν συχνά παράλληλα αυτές τις συνεδριάσεις. Θα συμμετάσχετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έλαβα κι εγώ μια απάντηση στο θέμα των πολωνικών λιμένων στα πλαίσια του σχεδίου αυτού. Euh, Για το θέμα της εφαρμογής ε, στην ε, Βαλτική, βεβαίως όλες οι υπηρεσίες εμπλέκονται, συνεργαζόμαστε, συντονιζόμαστε με τον Πατ Κόξ, με τους συναδέλφους, με όλους. Βέβαια ο καθένας ασχολείται με τα δικά του θέματα. Πάντως, κάνουμε συνεδριάσεις όπου συζητάμε όλοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Άρα λοιπόν στη πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης MOVE, ναι, ε, η συνεργασία είναι εξαιρετική. Πρέπει να σας πω πως και οι συγκεκριμένες περιφέρειες συντονίζονται και συζητάνε τα θέματα. Αυτό συνέβη και η Πολετονική Προεδρία και θα συμβεί η Πολανδική Προεδρία κυρίως και με όλους επόμενους, με την οποία ανταλλάξαμε απόψεις για το ποιος θα είναι ο συγκεκριμένος και αποφασιστικό ρόλος της ε, για τον διάδρομο αυτό. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη συνέπεια μεταξύ των όσων κάνουμε. Τώρα για το θέμα της Πολωνίας. Τα λιμάνια αυτά είναι σημεία τα οποία θα πρέπει να συνδεθούν και θα ήθελα η Πολωνία να προχωρήσει κάπως παραπάνω στο θέμα αυτό, γιατί η Γερμανία το έκανε για παράδειγμα για το Αμβούργο και για άλλα λιμάνια, το κάνανε οι κατοχώρες. Η Πολωνία βασίζεται πάρα πολύ στο εθνικό δίκτυο και στα interface που έχει. Είναι ένα περίπλοκο σύστημα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Πάντως για μένα τα πολωνικά λιμάνια θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη φιλοδοξία. Και το συζητήσαμε με την Υπουργό όταν τα είπαμε. Θα πάω εγώ στα πολωνικά λιμάνια για να συζητήσουμε το θέμα των στόχων και για το πώς βλέπουν αυτοί τα μελλοντικά του σχέδια. Ευχαριστώ. Έτσι κλείνουμε το θέμα της ημέρας της διάταξης. Κάθε, κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. So, wir kommen nun zum nächsten. θέμα Καλωσορίζω τον Κάρελ Βίνκ. Χρόνια τώρα, γνωστός μας, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής ε, Κίνησης. Γνωρίζει. Γνωρίζουμε ότι έχει 10.000 χιλιόμετρα δίκτυο, αλλά κανένας ε, όπου κανένας σειρμός δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Έχετε το λόγο κύριε Βίνκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω 10 λεπτά για να σας εξηγήσω ποια είναι η κατάσταση στο RTMS ή RTMS. Πολύ γρήγορα Πρέπει να δούμε αυτό το δίκτυο πώς μπορεί να ναι, γίνει ναι. διαλειτουργικό το σιδηροδρομικό δίκτυο. Όταν ξεκινήσαμε το 2005 είπαμε ότι ναι. Έχουμε λοιπόν την εναρμόνιση των λειτουργικών κανόνων, την χρήση τους, τους κανόνες δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αλλάξει και που πρέπει να ε, υλοποιηθούν αποτελεσματικά, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε κιόλα. Δέκα χρόνια τώρα έχουμε ξεκινήσει με την ε, ανάπτυξη των προδιαγραφών, την υλοποίηση των προδιαγραφών, την ε, θέση λειτουργία του ERTMS. Τώρα πρέπει να επιταχύνουμε, όπω είπαμε, και αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ένα πρόγραμμα ε, εισαγωγής ε, για το 2015-2016 χωρίς χρονοδιάγραμμα φυσικά δεν έχει κανένα νόημα άρα χρειάζεται το χρονοδιάγραμμα αυτό 2015-2016 για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα να ε, βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε την διαλειτουργικότητα στο δίκτυο με κύριες αρχές ότι μέχρι τώρα έχουμε δώσει πολύ χρόνο και προσοχή στο να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι προδιαγραφές και τώρα που έχουν οριμάσει πρέπει να μετακυλήσουμε την προσοχή μας προς τον χρήστη. Χρήστης σημαίνει και στη σιδηροδρομική επιχείρηση που πρέπει να είναι ανταγωνιστική και για λόγους περιβαλλοντικούς αλλά και για λόγους ε, ανταγωνισμού με, τις άλλες, με τους άλλους τρόπους των μεταφορών και για την αξιοποίησιμότητα, χρησιμότητα για τον ε, χρήστη το, ο μηχανισμός θα πρέπει να υπάρχει. Είπε ο πρόεδρος ότι έχουμε 10.000 ε, χιλιόμετρα, αλλά ένα σειρμός δεν μπορεί να το διατρέξει 10.000 χιλιόμετρα. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Τώρα με τους ε, επιτρόπους αλλά και με τους αρμόδιους για τη διαχείριση των υποδομών αλλά και με τον κλάδο πάνω απ' όλα προσπαθούμε να βρούμε μία λύση ώστε να έχουμε έναν σειρμό που μπορεί να διατρέξει τα 10.000 χιλιόμετρα ε, σιδηροδρομικής γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύσκολο έργο, δύσκολο καθήκον να τα καταφέρουμε. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε όλες τις ε, λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για τις υποδομές. Εστίαση βέβαια στις, ε, στην απασχόληση, Είχαμε την υποδομή, είχαμε τη βάση 1, τη βάση 2, τώρα έχουμε τη βάση 3 για τη διαλειτουργικότητα και τώρα προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη, διορθώνουμε, η ανάπτυξη των προδιαγραφών. Το ERTMS κοστίζει πολύ ακριβά. Οι προμηθευτές προσφέρουν υλικό σε επίπεδο υπερβολικά δαπανηρό, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Οι αλλαγές που χρειάζονται, και αυτό βέβαια είναι φυσιολογικό όταν ξεκινάει ένα σύστημα, Όλες οι αλλαγές αυτές που χρειάζονται λοιπόν κοστίζουν πολύ ακριβά για το χρήστη. Άρα με την τυποποίηση προσπαθούμε να μειώσουμε στο δυνατόν περισσότερο το κόστος. Για το πρόγραμμα Breakthrough 2015-2016 προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε σταθερά και όριμο σύνολο προδιαγραφών, διαλειτουργικέ διαλειτουργικές υποδομές, υποδομές που να τηρούν τις προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει τι, ε, ότι πρέπει να είναι και αυτές οι υποδομές σταθερές, να μην αλλάζουν ένα-δύο χρόνια, όπως σε κάθε αξιόλογο τέτοιο σύστημα. Πρέπει να έχουμε υπόψη όμως ότι ο χρόνος ζωής του τροχαίου υλικού είναι πολύ πιο μακρύς από το σύστημα και άρα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία με το χρήστη, σε συνεργασία με το χρήστη, ώστε να προβλέψουμε και την εξέλιξη των προδιαγραφών του ERTMS συν το χρόνο. Διαλειτουργικές λοιπόν και συμμορφούμενες υποδομές, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται δεκτή η μονάδα που χρησιμοποιούμε τώρα Πρέπει να δούμε πώς με τι χρονοδιάγραμμα και με τι προτεραιότητες θα κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και έτσι θα, θα προχωρήσει η συνεργασία και ο συντονισμός που έχουμε και με την άλλη συντονίστρια διότι εάν παραδείγματι πάρουμε την ε, ε, αλπική οδό ή την ε, μεσογειακή μπορεί να δούμε ότι υπάρχουν άλλες συνθήκες από αυτέ που επικρατούν σε άλλους, σε άλλους διαδρόμους άρα χρειάζεται ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Είχαμε αρχικά προσδιορίσει ως ε, σχέδιο το 2009 την πρώτη λύση για την ανάπτυξη, αλλά διαπιστώνουμε ότι δεν ήταν αρκετά ρεαλιστικό με την έννοια ότι δεν αντιστοιχούσε στις πραγματικότητες που αντιμετωπίζαμε. Και έτσι διατυπώνουμε μια διαφορετική ιδέα για το 2016 με ένα σχέδιο υλοποίησης του ERTMS σε υποδομές προκειμένου να έχουμε πιο διαλειτουργικό δίκτυο. Διευκόλυνση της ανάπτυξης, ε, μάλλον καλύτερα ε, καθαρό και διαφανές ε, σύνολο κανόνων. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Χρειάζεται να υπάρχουν διαφανή ε, διαφανείς κανόνες, διαφανές πλαίσιο κανόνων. Είναι πολύ περίπλοκη αυτή τη στιγμή η εικόνα που δίνει ένα περίπλοκο πλέγμα εθνικών διατάξεων και άλλων και βεβαίως δεν θέλουμε να ε, καταργήσουμε τις διατάξεις. Θέλουμε όμως να κάνουμε ένα χτένισμα, ένα ξεκαθάρισμα αυτού του συστήματος ώστε το ERTMS να μπορεί να υλοποιείται παντού. Διευκόλυνση της ανάπτυξη το ανέφερε η Κατρίν ισχύει για κάθε διάδρομο. Και οπωσδήποτε για τις επενδύσεις που χρειάζονται για το ERTMS. Συγχρηματοδότηση με το ΣΕΦ και άλλα μέσα βεβαίως ε, με επιχειρηματικά επιχειρήματα ε, και το λέω αυτό ιδιαίτερα γιατί αυτό που δεν κάναμε και αυτό που δεν λαμβάνουν υπόψη οι επιχειρήσεις είναι ότι υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή δεν εξυπηρετούν μόνο την ασφάλεια οι επενδύσεις αυτές ή την, ε, τις ανάγκες εξυπηρέτησης του κοινού. Πρέπει να κοιτάξουμε και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και τις συνθήκες ασφαλείας και το κόστος και τη μείωση σε κατανάλωση ενέργειας. Όλα αυτά είναι ένα σύνολο επιχειρηματολογίας για την ε, εξυπηρέτηση μιας επένδυσης που πρέπει να προβάλλουμε για το ERTMS. Ρεαλιστική και αποφασιστική ανάπτυξη μέσα από σχέδιο που αναπτύσσεται σε δύο σχέδια, σε δύο βήματα, όπως συμφώνησαν τα κράτη-μέλη άλλωστε. Πρώτα από το 2015 στο 2020 και μετά η δεύτερη περίοδος 2020. 2030 η πρώτη φάση ολοκληρώνεται το 2015. Τελειοποιείται καλύτερα το 2015, όπου θα έχουμε την αναθεωρημένη έκδοση και τις ανάγκες σε διαλειτουργικότητα και το δεύτερο βήμα, όπως είπαμε, θα εκτελεστεί από το Σεπτέμβριο 2015 έως τον Απρίλιο 2016 με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υλοποίησης μέχρι το Απρίλιο του 2016 και τα σχέδια τα οποία σας ανέφερα και τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα. Συνεργαζόμαστε με κράτη-μέλη, με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατά τρόπο αγαστό και πέραν των συνεδριάσεων που ήδη υπάρχουν έχουμε εισαγάγει τριμερείς όπως τις ονομάζω επαφές με ε, ηγετικά στελέχη πολιτικών ε, υπουργείων, επασφερτώσει, πολιτικών αρχών, ε, με υποδομές, με διαχείριση υποδομών, με επιχειρήσεις δρομικές, όπου κοιτάμε πού βρίσκονται οι στενοποί, λαμβάνουμε τις σχετικές αποφάσεις και αυτό έχει να κάνει με θέματα όχι μόνο τεχνικά, αλλά και με οικονομικές δυνατότητες. Αφού είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο των Οικονομικών των Πρώτων Μελών. Άρα, αν κοιτάξουμε ε, το 2016 έως το τέλος του 2016 θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης με καλύτερη απεικόνηση αλλά και πιθανολόγηση για την υλοποίηση των στόχων μας ώστε να έχουμε διαλειτουργικό δίκτυο σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2016. Είναι πολύ σημαντικό σχέδιο, είναι το πιο προηγμένο, το πιο προχωρημένο ως προς την υλοποίηση και τον ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για διάφορα έργα, ιδίως υποδομών, ώστε να υποστηρίξει και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το σχέδιο είναι έτοιμο, τεχνικά είμαστε έτοιμοι. Η δε υποστήριξη μας προσφέρει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, όλοι αυτοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε, αποτελούν νομίζω την καλύτερη εγγύηση να επιτύχουμε τον κύριο στόχο, στόχο μας. Ευρωπαϊκή Ένωση διαλειτουργική στους σιδηροδρόμους. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Κουν, τρικέ, υποφαινόμενος, έτερος. Τέλτσκα. Δύο λεπτά ο καθένας, ό,τι και να είναι. Κουλ. Cool. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ το συντονιστή. Κάρελ Βίνκ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα ζητήματα της ασφάλειας. Ε, η αποφυγή ατυχημάτων και επεισοδίων, η ασφάλεια των επιβατών. Θυμάμαι ότι είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε με πολύ μεγάλη έμφαση συζητήσει ε, στις Βρυξέλλες, γιατί είχαμε μεγάλο αριθμό ε, ατυχημάτων πριν από μερικά χρόνια, ε, με πολλά θύματα, όταν δεν είχαμε, επί παραδείγματι, τήρηση των συνθήκων ε, πέδησης, όταν άναβε το κόκκινο φορνάρι ή εάν έπρεπε να σταματήσει το τρένο ευνηδίως γιατί βρισκόταν κάποιος πεζός πάνω στην ε, Ράγα. Είναι ζητήματα τα οποία έχουμε συζητήσει, είναι ζητήματα τα οποία, στα οποία έχουμε την, τονίσει το πόσο ε, κατεπήγον είναι να προχωρήσουμε σε συνθήκες ασφαλείας και είπε ο εορτάζων πρόεδρος ότι έχουμε μεγάλες γραμμές, γραμμές μεγάλες ταχύτητας που καλύπτουν και την τοπική και την περιφερειακή κυκλοφορία. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι με να λειτουργεί όλο αυτό το δίκτυο με ένα σύστημα INTS e που θα ε, ε, μεταδίδει συντονισμένα τα σήματα κινδύνου ασφαλείας ανεξαρτός σύνορων. Αυτό θα είναι το καθοριστικό. Η τρίτη μεγάλη ε, πάροχη συστημάτων, η Alstrom, η Dominique Alstrom, η Bombardier και η Siemens, αντίστοιχα Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, δεν έχουν προσφέρει ένα νέο σύστημα για να μπορεί να λειτουργήσει με το EMTS ένα σύστημα ασφαλείας. Και ρωτώ, Κάρελ, έχεις κάποια παραδείγματα που να μας δείχνουν ότι λειτουργεί το σύστημα πέραν των εθνικών συνόρων με το ICE, ε, το Διεθνές Γρήγορο Τρένο το Γερμανικό. Μπορεί να πάει ε, μέχρι το Παρίσι από τη Γερμανία ή μέχρι την Πολωνία. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις καθυστερήσεις, ε, διαταραχές ε, στο, στην κυκλοφορία λόγω προβλημάτων των σημάτων. Αυτή είναι η δουλειά σας. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, μαζί με τους τρεις παρόχους συστήματος όπως έλεγα. Αυτά. Και βέβαια θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με μεγάλη έμφαση. Ντομινίκη Κρικέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κάριλ Βίνκ για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχω τέσσερις ερωτήσεις. Καταρχήν, τι πιστεύετε για τη θέση του Συμβουλίου για το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους στο τεχνικό φάκελο που προσπαθεί να αποκεντρώσει κατά κάποιο τρόπο τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Σιδηροδρομικής Αρχής ε, έχοντας αρχές τερματικών σταθμών που θα αναλάβουν την ευρωπαϊκή διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου. Εδώ δεν μιλάμε για ενοποίηση αλλά για εκ νέου εθνικοποίηση. Δεύτερον, ποια είναι η σχέση μεταξύ της στήριξης επενδύσεις από την Ευρώπη και πώς αυτό θα επηρεάσει τις υποδομές και πώς σχετίζεται αυτό με την ανάγκη να έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή διαχείριση στις υποδομές που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη. Τρίτον, τι πιστεύετε για μια πρόταση που έχει κατατεθεί για να έχουμε μόνο μία κοινή χρηματοδότηση και ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη με το συγκεκριμένο μηχανισμό που έχει προταθεί. Και τέλος, ποια θα είναι η οικονομική απόδοση αυτού του ευρωπαϊκού ε, μηχανισμού διαχείρισης για τους σιδηροδρόμους. Υπάρχει κάποιος, ε, κάποια τέτοια δυνατότητα, δηλαδή να έχουμε και μια οικονομική διάσταση ε, και ένα τμήμα βεβαίως των εσόδων θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη-μέλη σύμφωνα με μια κλίδα κατανομής που μένει να αποφασιστεί. Επίσης και άλλη μια ερώτηση. Πώς μπορούμε το σύστημα αυτό να το εξαπλώσουμε και εκτός Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Λέω κύριο Στελίτσκα. Ήταν πολύ σαφής η παρουσίαση και μπορώ να συνταχθώ με τους ε, στόχους και τις στρατηγικές ε, σημασίας προσπάθειες που γίνονται. Νομίζω πως όλοι εδώ στην αίθουσα καταλαβαίνουμε πως τη συμφόρηση την προκαλεί η χρηματοδότηση. Και χαίρομαι που αναφερθήκατε σε κάτι στο οποίο είχα σκοπό να σταθώ. Νομιμοποιείται ε, η δημιουργία ενός business plan γιατί είπατε πως θα ασχοληθείτε με το θέμα αυτό και ίσως θα έπρεπε να το έχουν τονίσει προς τα κράτη-μέλη εδώ και καιρό. Δηλαδή, για το άμεσο μέλλον, τι θα γίνει έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να καταλάβουν ακριβώς ότι τι γίνεται, το ότι υπάρχει επιχειρηματική προοπτική ε, και ότι υπάρχει επιχειρηματικό μοντέλο που θα πρέπει στο σύστημα αυτό το ευρωπαϊκό που στείλουμε να ε, απηχείται. Τώρα θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια. Τα πλεονεκτήματα να έχουμε τουλάχιστον 20% καλύτερη αξιοποίηση των υφισταμένων ε, γραμμών. Δεύτερον, η ασφάλεια. Και τρίτον, το κόστος. Εάν δεν χρειάζεται να ε, παράγονται διαφορετικοί σειρμοί για, για το κάθε κράτος μέλος, προφανώς και μειώνεται σημαντικά το κόστος και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να προβληθεί και το πλεονέκτημα, το οικονομικό. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων θα έχει την τελευταία λέξη, αλλά όταν έχουν γίνει τόσα λάθη εδώ και, 7, τόσα χρόνια και έχουν δαπανηθεί και κατασπαλταληθεί τόσα χρήματα, πρέπει τα κράτη εν τέλει να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης. Κάπως πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Και επίσης για τα επόμενα 15 χρόνια είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι δεν θέλουν να γίνει καμία αλλαγή και να μην γίνει καμιά ανταλλαγή απόψεων με τις ε, υπηρεσίες της Επιτροπής και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων. Δηλαδή έχουμε κλείσει τα επόμενα 15 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Πρέπει να υπάρξει κάποια παρέμβαση και αν υπάρχει κάποια τεχνολογική εξέλιξη που ασφαλώς και θα προκύψει τα επόμενα 15 χρόνια, πρέπει αυτή να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ε, ότι είναι συμβατή. Το είχαμε δει και στο παρελθόν. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ένα συμβασμό, χωρίς να χρειάζεται να τροποποιηθεί κάθε δυνατή σύμβαση, αλλά να είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και μια τελευταία ερώτηση. Είχατε πει ότι, είναι δυνατότητα, ότι υπάρχει δυνατότητα συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 50% του ERTMS. Υπάρχει λοιπόν η συγχρηματοδότηση αυτή και σε ποια κατεύθυνση βαίνει. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε προχωρούν διάφορα σχέδια. Υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα επαναληφθούν τα ασφάλματα των, προηγουμένων δεκαετών στο μέλλον. Ναι, Πρόεδρε, και εγώ θα προσθέσω κάτι. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των εισαγωγών σειρμών τροχαίου υλικού από ξένες, από τρίτες χώρες, κινέζικα κτλ. Και πώς κρίνεται το θέμα της συμβατότητας εν προκειμένου. Ναι, μα ούτω ή άλλω όμω, λέει ο πρόεδρο, αυτό το σύστημα υπάρχει και το έχουν υιοθετήσει ε, και πολλά κράτη εκτό Ευρώπη. Εμεί μπορεί να το εφήβραμε, αλλά οι άλλοι το έχουν υιοθετήσει με μεγάλο ενθουσιασμό. Uh, πρώτα πρώτα θα ήθελα να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Προτίθεκα τι γίνεται με τους προμηθευτές, τι πολιτική υπάρχει, τι, τι προσδοκίες υπάρχουν. Κοιτάξτε, η βιομηχανία και το έχω συζητήσει με τα κορυφαία στελέχη, θα το πούμε και στη Ρίγα. Αλλάζει, αλλάζει δομικά, διαρθρωτικά πάρα πολύ. Τελευταίο εξάμεινο με την ε, εξαγορά της Ανσάλτο από την Ιχιτάτσι Μπαίνουν τώρα οι Κινέζοι στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται να διαδραματίσουν ρόλο οι προμηθευτές οι Ασιάτες. Επίσης για τους ε, Ευρωπαίους προμηθευτές έχουμε κάποια υλικά που προέρχονται από την Χιτάτσιο και αυτά τα υλικά είναι το ίδιο καλά με τα ευρωπαϊκά, αν όχι καλύτερα. Οπότε και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των βιομηχανικών περιοχών, ότι ε, έχουμε προϊόντα πάρα πολύ καλά πλευρά χρήστη, ε, γενική, αλλά δεν μπορούμε αυτό να τα θέσουμε σε εμπορία. Γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη αρκετά ποιοι είναι οι χρήστες. Οπότε οι Ζήμες και οι με αυτό τώρα νοιάζονται. Με αυτό τώρα ασχολούνται. Και αυτό και θα συζητηθεί στη συνάντηση τη Τώρα, όσον αφορά τα διασυνοριακά, ρωτήσατε. Το, το, το, το σημείο διέλευση των σύνορων υπάρχουν ε, ε χώρες ε, που υπάρχει αυτό έχει καθοριστεί α πούμε Βέλγιο Ολλανδία και έχει κοστίσει πολύ σε χρόνο και χρήμα αλλά έτσι είναι το ζήτημα είναι βέβαια ότι το εξετάζουμε στα πλαίσια αυτού του πρωτοπόρου προγράμματος Έτσι γίνεται η ανάλυση του διασυνοριακού παράγοντα που εάν επιληθεί θα επιληθούν και άλλα μαζί. Τα τεχνικά προβλήματα της συμβατότητα τη υποδομή, το πρόβλημα εγκρίσεων και αδειών, οπότε κάθε διασυνοριακή διέλευση θα πρέπει να αποτελέσει ένα έργο και έτσι να εξεταστεί. Αυτό το κάνουμε τώρα επίσης. Επίση συζήτησα και με κάποια κράτη-μέλη. Όχι όλα, με κάποια κρατημέλη για να αποφασίσουμε ποιε είναι οι προτεραιότητε όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων. Α πούμε, Γερμανία. Έχουμε 12 τέτοια σημεία. Και σε συνεργασία λοιπόν με του διαχειριστέ ε, τη υποδομή και με το Υπουργείο είπαμε ότι 2015-2020 θα δώσουμε προτεραιότητα σε πέντε τέτοια σημεία από τα 12. Τα πιο σημαντικά από πλευρά ε, ε κυκλοφορία, από πλευρά κίνηση από την όμορφη χώρα ή τι όμορφε χώρε. Εδώ είναι η προτεραιότητα γιατί πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνει τώρα. Άλλη ερώτηση του κ. Ρίκε. Ήδη είπαμε ε, για τη σχέση αυτών που συζητούμε τώρα με το τέταρτο πακέτο για και θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια πολύ γερή προσπάθεια συντονισμού από τις ε, υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν σε επίπεδο κρατών μελών. Οπότε θα πρέπει επίσης να γίνει κάποιο είδους αναθεώρηση, χτένισμα της νομοθεσίας, ούτως ώστε η νομοθεσία για τη διαχείριση των δρόμων και του ευρωπαϊκού συστήματος να μην είναι φραγμός. Τώρα, για τις νέες υποδομές. Οπωσδήποτε θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε τι ισχύει για το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης δρόμων. Για την χρηματοδότηση τώρα. Κάτι το οποίο το ρώτησε ο κύριος Ρικέ και ο Πάβελ, είναι θέμα νοοτροπίας στους ιοδρόμους. Όταν χρειάζεται χρηματοδότηση, τότε για υποδομές, για κάποιο έργο, πάνε και ζητάνε χρήματα από την κυβέρνηση. Οπότε για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης. Εδώ να δούμε τι θα απογίνει η επένδυση. Δυνατότητες, ασφάλεια, ε, κατανάλωση ενέργειας, όλες αυτές οι μεταβλητές αντιπροσωπεύουν κόστος. Οπότε υπάρχει εδώ κάποια θετική επιρροή απλώς κόστους για την εμπόρικη αυτή προσπάθεια. Και κατόπιν βλέπουμε ποια είναι η απόδοση και να δούμε μετά τι πολιτική υπάρχει όσον αφορά την πρόσβαση στην υποδομή. Πώς θα τα λύσουμε αυτά, πώς θα έχουμε ένα ισορροπημένο σύστημα, γιατί έχουμε μεγάλες διαφορές από κράτος σε κράτος. Οπότε το εισόδημα, η απόδοση δεν έχει ληφθεί ακόμη υπόψη για την ε, κάθε ε, ε, απόπειρα του επιχειρήν. Οπότε έτσι θα κρυφθούν αυτέ οι επενδύσει. Τώρα, όσον αφορά την αναπτυξή μα εκτό Ευρώπης, υπάρχουν πολλά προγράμματα και σχέδια τα οποία γίνονται εκτό Ευρώπη. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα του σημείου διάβαση των συνόρων. Γίνεται σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Άρα αυτή την άποψη δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, αν εκεί, ε, ε, εδώ, μάλλον εδώ στην Ευρώπη, έχουμε αυτό το πρόβλημα της διάβασης των συνόρων. Άρα, αν εδώ πέρα δοθεί μια λύση και αποκτήσουμε αυτή την εμπειρία, αυτό είναι τεχνολογικό πλεονέκτημα. Έτσι, επομένω, θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τις επιχειρήσεις μας. Επίσης, μιλάμε για την τεχνολογία τώρα. Στο σημείο βρισκόμαστε τώρα. Και επιδέχεται ανάπτυξη αυτή η τεχνολογία. Βέβαια σε 10-15 χρόνια μπορεί να έχουμε άμεση σύνδεση με έναν δορυφόρο αμέσω του συστήματος του Γαλιλαίου. Οπότε δεν χρειάζεται τίποτα πια όσον αφορά την υποδομή. Όλα θα συνδέονται με άμεση σύνδεση ε, από το δορυφόρο στο έδαφος. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα επιδέχεται ανάπτυξη, επιδέχεται εξέλιξε αυτή η τεχνολογία. Fink, thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Και ελπίζουμε ότι θα διδαχθούμε από τα σφάλματα και θα είναι καλύτερο το μέλλον από το παρελθόν. Συνεχίζουμε με την επόμενη συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών στον μόνο.